I have already uh, introduced Ήδη σας ε, σύστησα, θα σας ξαναπαρουσιάσω. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ε, ευρωεκλογές. Ε, τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες. Για πείτε μας. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε. Με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ. Είσαστε αρκετοί. Βλέπω με χαρά ότι το θέμα σας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει τους ε, δημοσιογράφους. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να σας ικανοποιήσει το σεμινάριο. Θα μιλήσουμε για τις ευρωεκλογέ και για το πώς θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για τις γυναίκες και τα θέματα των γυναικών. Για να δούμε πού έχουμε φτάσει καταρχήν. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί και αν δεν το ξέρετε σας το λέω, να εξαλείψει την ισο... τις ανισότητες και να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές του. Το 1957 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνθήκη της Ρώμης προβλεπόταν η αρχή ότι τα δύο φύλλα θα πρέπει να αμείβονται το ίδιο για την ίδια εργασία. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα πρώτο βήμα ένα απαραίτητο βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Την επόμενη δεκαετία αυτό έφτασε σε πολλούς τομείς όπου η μεταχείριση δεν ήταν ισότιμη για τα δύο φύλλα. Παραδείγματα, η πρόσβαση στην εργασία, κατάρτιση, οι προαγωγές, συνθήκες εργασίας, ίσο μισθό και κοινωνική ασφάλιση, δικαίωμα στη γονική άδεια, παραβίαση και βία εναντίον των γυναικών κτλ. κτλ. Πολλά νομοθετήματα υιοθετήθηκαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε τώρα όμως παρά τα βήματα που έχουμε κάνει να πάμε ακόμα παραπέρα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Βία εναντίον των γυναικών. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπομορφή έμφυλη διάκρισης. Διάκριση δηλαδή λόγω φύλου. Την περασμένη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία για τα δικαιώματα των γυναικών ε, από την ε, Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε σε μία επίσκεψη στην Μαδρίτη, στην ε, χώρα μου, για να δει επιτόπου τι προσπάθειες έχει κάνει η Ισπανία για να καταπολεμήσει την βία κατά των γυναικών στο εσωτερικό της χώρας. Η αντιπροσωπεία βρήκε ότι η Ισπανία έχει θέσει το τον πύχη για όλα τα κράτη-μέλη, για τον τρόπο με τον οποίο ε, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτή τη βία λόγω φύλου. Σήμερα Δυστυχώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Η υγεία και η εκπαίδευση είναι τομείς όπου υπάρχει μεγάλη βελτίωση, η απασχόληση, η πρόσβαση στην, ε, σε οικονομικούς πόρους και οι ηγετικές θέσεις είναι τομείς όπου οι γυναίκες ειστερούν. Ε, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε ισότητα ανδρών και γυναικών. Με βάση το τελευταίο ευρωβαρόμετρο για το θέμα αυτό, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η προώθηση τη ισότητα των φύλων είναι σημαντικό θέμα για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία. Το πιστεύουν το 91% των Ευρωπαίων για την οικονομία, το 87% των Ευρωπαίων το πιστεύει ή απλώ για αυτού προσωπικά είναι σημαντικό. Το 84% πιστεύει ότι είναι προσωπικά για αυτού σημαντικό. Το, σημαντικό, το σημερινό θέμα είναι οι γυναίκες στην πολιτική. Η ίση συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων σε όλους τους τομείς ε, των αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλής διακυβέρνησης. Από τις 20 ε, χώρες παγκοσμίω με τον υψηλότερο ε, ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, οι 6 είναι ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Όμως, Τρεις από, τις, ε, τρεις από τους 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι γυναίκες στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Λιθουανία. Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπούνται στην ε, κυβέρνηση και στις ανώτερες θέσεις στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή το 37% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γυναίκες σε σχέση με το 27,9% που έχουν τα κράτη-μέλη στα εθνικά τους κοινοβούλια, κατά όρο. Ακούσατε προηγουμένως την Virginia Langback, που είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που σας μίλησε για την έλλειψη ισορροπίας στην εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Και πάω κατευθείαν στο θέμα για το οποίο ήρθα να σας μιλήσω, τις ευρωεκλογές και τι κερδίζουν οι γυναίκες τις ευρωεκλογέ. Και ποια είναι η διαφορά που θα κάνει η ψήφος των γυναικών, αν πάνε δηλαδή οι γυναίκες να ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωεκλογέ, τι θα πετύχουμε. Μένουν λιγότερο από τρει μήνε για τι ευρωεκλογέ που θα γίνουν από τι 23 έω τι 26 Μαου. Οι Ευρωπαίοι πολίτε με τι επιλογέ του θα διαμορφώσουν τις, την καθημερινότητά του και την καθημερινότητα των οικογενειών του, την Ευρώπη και τη χώρα τους ή τη χώρα που, στην οποία θέλουν να ζήσουν. Είναι μία από τις πιο αποφασιστικές εκλογές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ που είναι προβληματικές δεν είναι εύκολες. Η Ρωσία, οι προβλήματα παραπληροφόρησης, fake news, ε, ψευδείς ειδήσει για τις εκλογές, λαϊκισμός, εξτρεμισμός, όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πάνω από μια δεκαετία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι εκλογείς θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της χώρας τους ε, που θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιο θα είναι, με την, θα αποφασίσουν δηλαδή με την ψήφο του, ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γυναίκε είναι πολύ δυνατές σε νούμερα, δηλαδή έχουν μια ισχυρή ψήφο. Το 2017 είχαμε 104,6 γυναίκες για 100 άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η αναλογία με βάση τα νούμερα της Eurostat. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για να προχωρήσουμε, για να εξασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων και να δώσουμε μεγαλύτερη εξουσία στις γυναίκες ψηφίζοντας για εκπροσώπους που είναι υπέρ της ισότητας των φύλων και που θα περάσουν νομοθεσία ε, για δίκαιη μεταχείριση, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέτουν τους όρους για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία που θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Εάν ψηφίσετε για έναν εκπρόσωπο που θα σας εκπροσωπήσει εσάς και τα συμφέροντά σας, θα διαμορφωθεί μια ατζέντα ισότητας για ένα ισότιμο μέλλον. Με βάση τις ε, σφιγμομετρήσεις πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τεράστιο κατακαιρματισμό μετά τις επόμενες εκλογές. Θα ανέβουν τα λαϊκιστικά και ακραία κόμματα. Για πρώτη φορά από τις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές που έγιναν το 1979, τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, οι δύο μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές, μπορεί να μην φτάσουν στην ε, απαραίτητη πλειοψηφία για να μπορούν να περνάνε νομοθεσία και να κάνουν συμφωνίες. Το μείγμα λαϊκιστών και ακραίων κομμάτων δεν είναι πιθανό σε αυτή τη φάση να είναι αρκετά δυνατό για να αντιστρέψει την πρόοδο που έχουμε επιτύχει για την ισότητα των φύλων. Αλλά, υπάρχει πάντα ένα αλλά, θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό το μείγμα ένα εμπόδιο για να μην υπάρξει περαιτέρω ε, πρόοδος. Γιατί υπάρχουν φωνέ που ακούγονται ότι έχουμε αρκετή ισότητα φίλων ή το έχουμε παρακάνει και με την ισότητα των φίλων. Και τώρα φτάνω στο τέλο τη παρεμβασή μου. Θα ήθελα να σα τονίσω ακόμα μια φορά τη σημασία αυτών των ευρωεκλογών για εσά. Εγώ πιστεύω ότι είσαστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι και φιλοευρωπαίοι και θα πρέπει να δίνετε σημασία στην αξία της ε, δημοκρατικής ε, συμμετοχής και να καταλάβετε τις ε, συνέπειες του να ψηφίσετε ή του να μην ψηφίσετε. Ευχαριστώ. Θα δεχθεί κάποιες ερωτήσεις ο κύριος Καρμόνα πριν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Σηκώστε τα χέρια λοιπόν. Όχι, ε, δεν θέλετε. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Πριν φτάσετε Είχε γίνει μια ερώτηση από την αίθουσα ε, για το ενδεχόμενο ε, εναλλαγής, εκπεριτροπής ε, ορισμού δηλαδή των πρόεδρων του Κοινοβούλου. Δεν είστε ε, ίσως αρμόδιος, αλλά τέλος πάντων ε, το θέμα ήταν πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες ε, εδώ στην ηγεσία, στο πιδάλιο του Ευρωκοινοβουλίου. Ήταν μόνο δύο μέχρι τώρα οι γυναίκες πρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου. Έχει ποτέ προκύψει αυτό στη συζήτηση, το έχετε αναφέρει στο πλαίσιο των συζήτησεων για το οργανόγραμμα. Τι θα μπορούσε να γίνει, ίσω και ποια είναι προ τον κρατών μελών ενδεχομένω, αν έχετε να πείτε κάτι. Απάντηση. Ακούστε, το βασικό εδώ είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν θα ψηφίσετε για κάποιον που θα έρθει εδώ για να παρασπίσει τα δικαιώματα των γυναικών. Αν γίνει αυτό, άμεσο αποτέλεσμα θα έχει να έχουμε περισσότερες γυναίκες στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ψηφίσετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επηρεάσετε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο, την ευρωπαϊκή ατζέντα. Άπαξ και γνωρίζουμε τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών σε ό,τι αφορά τα διάφορα αξιώματα. Ο ορισμός σε αυτά θα γίνει με βάση και το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αλλά θα έχει γίνει ήδη η επιλογή. Θα έχουν δηλαδή προωθηθεί ε, τα θέματα ισότητας του φύλου. Άρα τώρα είναι η στιγμή να μπουν στην ατζέντα τα θέματα της ισότητας των φίλων Και με την ψήφο σας μπορείτε να επηρεάσετε. Γιατί το μετά θα εξαρτηθεί κατά πολύ από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ερώτηση. Είπατε ότι μας μένουν λίγο πολύ τρεις μήνες. Είστε και επικεφαλής ε, του τμήματος για τον τύπο. Εσείς πώς έχετε σκεφτεί ε, να στοχεύσετε στις ε, γυναίκες. Είπατε 104 και κάτι γυναίκες ε, έναντι 100 ανδρών, άρα είναι πολλές οι γυναίκες οι ψηφοφόροι που θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Τι έχετε προβλέψει, απάντηση. Εμείς εστιάζουμε στη σημασία που έχει να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές αξίες. Όλα αυτά που κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο έχει αυτή τη στιγμή, είναι ο μεγαλύτερος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Και βέβαια εδώ περιλαμβάνουμε και την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, μη διακριτική μεταχείριση. Άρα η ισότητα των και γυναικών φυσικά και έχει εξέχοντα ρόλο και εξέχουσα θέση. Σε εσά που κατά κάποιο τρόπο είστε μας, πάντοτε σας υπενθυμίζουμε τη σημασία που έχει. Να πάει κανείς να ψηφίσει κόμματα τα οποία προασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί αυτόματα το αποτέλεσμα θα είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων σας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αν, γιατί ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία, το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα τα ευρωπαϊκά είναι πολύ ψηλό εκεί. είναι από τις χώρες που είναι πιο ψηλά. Όμως, σε ό,τι αφορά την προσέλευση στις κάλπες για τις ευρωεκλογέ, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά εκεί. Άρα, εσείς θα πρέπει να περάσετε το μήνυμα. Γιατί δεν θα πρέπει μετά να σας εκπλήξει αρνητικά το ότι αυτοί που εξελέγησαν βουλευτές και κόμματα δεν είναι αυτοί που προασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες και τα συμφέροντα των χωρών σας. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα. Ενημερώστε παρακαλώ τους ψηφοφόρους. Ενημερώστε τους πολίτες για το πόσο σημασία έχει να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Εσείς με το κίτρινο. Πρέπει να πιστέψουμε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες δεν ψηφίζουν αρκετά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες ψηφοφόροι ή το μείγμα. Δηλαδή τι ε, τους δίνουμε εμείς ως πληροφορίες είναι το πρόβλημα. Γιατί οι γυναίκες έχουμε σε κόμματα εξτρεμιστικά ή ευρωσκεπτικιστικά. Ε, έχουμε το κόμμα τη Μαρή Λεπέν, για παράδειγμα, να το ξεχνάμε αυτό. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι, πώ ενημερώνουμε τις γυναίκες. Τι κίνητρα τους δίνουμε ή ότι δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκες. Απάντηση. Είναι λίγο πολύ όλα όσα είπατε. Το ότι δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκε ψηφοφόροι σίγουρα είναι ένα θέμα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στι εκλογέ, τα νούμερα που έχουμε δείχνουν ότι είναι λίγο πολύ 50-50. Άρα διάκριση δεν υπάρχει εκεί, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, ε, αυτοί που πάνε να ψηφίσουν είναι λίγο πολύ κατά 5% κατά 5% γυναίκες. Αυτό όμως που εμένα με εντυπωσίασε και με ξέπληξε, προετοιμάζομενος για αυτή την ε, ε, Συνεδριάστηκαν κάποια στοιχεία που διάβασα από την εξωτερική υπηρεσία ε, έρευνας του ε, Κοινοβουλίου. Είδα λοιπόν ότι υπάρχουν χώρες που πραγματικά υποεκπροσωπούνται. Οι γυναίκες εκεί, στην κυβέρνηση, σε εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι λοιπόν όταν, όταν αυτές οι γυναίκες, το 5% πάνε να ψηφίσουν, τις εθνικές ευρωεκλογές, τοπικές εκλογές. Μήπω για αυτέ δεν είναι θέμα κλειδί το θέμα τη ισότητα των δύο γιατί αλλιώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ. Για παράδειγμα, στι χώρε που είναι στην κορυφή, δηλαδή που έχουν τι περισσότερε γυναίκε εθνικέ κυβερνήσει, εθνικά κοινοβούλια, που είναι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Και Ουγγαρία που έχει τόσες λίγες γυναίκες σε μεγάλα έτσι, ψηλά αξιώματα μαζί με τη Μάλτα. Γιατί είναι τόσο τεράστιο αυτό το χάσμα. Δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει. Τι κάνουμε για τις γυναίκες αυτές. Γιατί δεν τις παροτρύνουμε να ψηφίσουν κόμματα που υποστηρίζουν τις ευκαιρίες και την ισότητα των φίλων η Ιταλίδα εκεί, ρεπόρτερ. Σε σχέση με τη στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης, μιλάω για τη δική μου χώρα, την Ιταλία, που υπάρχει μεγάλη καχυποψία αυτή τη στιγμή από τον κόσμο στα παραδοσιακά μίντια. Ό,τι γράψουμε λοιπόν εγώ και στη δημοσιογράφη, οι συνάδελφοί μου, δεν νομίζω ότι θα γύρει την πλάστιγκα υπέρ ε, της ε, ψήφιση περισσότερων γυναικών. Ε, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες στρατηγικές για να διεισδύσουμε στο εκλογικό σώμα που δεν διαβάζει ή δεν ε, ακούει παραδοσιακά μέσα αλλά να ζητεί στο ίντερνετ τα πληροφορίες και ενδεχομένως να παραπλανάτε ή να παραπληροφορείτε από τις ψευδείς ειδήσει. Καλή ερώτηση. Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσει είναι κάτι που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε στην εκλογική αυτή εκστρατεία, διότι πραγματικά το βλέπουμε το πρόβλημα. Τώρα που πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ. Και μάλιστα αυξάνει το φαινόμενο. Θέλω να πω πως αυτά που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τις ψευδείς ειδήσει και την παραπληροφόρηση είναι ότι δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τις ψευδείς ειδήσει και την παραπληροφόρηση είναι να αποσταθεροποιήσουν το δημοκρατικό μας σύστημα. Πολύ παραπληροφόρηση έρχεται, για παράδειγμα, από τη Ρωσία με αυτό το σκοπό. Δεν θέλω να μπω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες γιατί δεν είναι και το αντικείμενο του σεμιναρίου σήμερα, αλλά έχουμε πολύ πρόσφατα στην επικοινωνική μας στρατηγική συγκροτήσει μια ειδική μονάδα που θα ασχολείται με ακριβώς αυτές τις εκστρατείες παραπληροφόρησης. Προσπαθούμε λοιπόν να αναζητήσουμε ψευδείς ειδήσει. Δεν βλέπουμε να κυριαρχεί το θέμα της σώτας των φίλων. Ναι, αλλά έχετε μια ειδική στρατηγική ε, ενημέρωσης, πληροφόρησης. Ένα είναι πώς κανείς ε, θα καταρρύψει τις ψευδείς αλλά εγώ μιλάω για μια στρατηγική που μπορεί να έχετε ενδεχομένως ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενημερώσετε τους πολίτες για το τι συμβαίνει. Κύριο στον συνήθως τα κόμματα που διαδίδουν ε, ψευδείς ειδήσει ε, είναι πολύ κακά για τις γυναίκες κατά μέσο It's a question or a comment, I <laughs> No, Ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, ερώτηση. Έχετε κάποια θετική στρατηγική ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, υπάρχει μια στρατηγική δική μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια, ένα από τα στοιχεία είναι να κάνουμε αυτά τα σεμινάρια. Είναι τμήμα της στρατηγική μας για να περάσουμε μηνύματα μέσω των δικών μας μέσων ενημέρωση για ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε της. Μερικές φορές, όταν ο πολίτης ρωτάει γιατί πρέπει να ψηφίσω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να κατέβουν στη γη, πρέπει να προσγειωθούν. Ε, και πρέπει και το Κοινοβούλιο να ε, προσγειωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσγειωθεί για να κάνει πράγματα για αυτούς. Έχουμε μία app, μία εφαρμογή που έχουμε ε, αναπτύξει για το τι κάνει η Ευρώπη για σένα. Έτσι τη λέμε αυτή την εφαρμογή. Έχουμε μία σειρά από δελτία που εξηγούν σε κάθε κοινωνική ομάδα ποια είναι η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της χώρας, από τη συμμετοχή τη χώρα τους στην Ευρώπη. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τα ίσα δικαιώματα. Υπάρχουν ειδικά δελτία με πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τα δικαιώματα ε, των ΛΟΑΔΑ για να καταπολεμήσει τον διαβήτη, ε, για την υγεία δηλαδή, πακέτα ενημερωτικά, διαβάστε τα, σας καλώ να τα διαβάσετε, γιατί έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα εκεί που θα σας βοηθήσουν εν ώψη των ευρωεκλογών. Μία τελική ερώτηση παρακαλώ θέλω να ακούσω. Μόνο. Παρακαλώ. Μπορείτε να μιλήσετε και ελληνικά για τα fake news, για τις ψευδείς ειδήσει που άκουσα από, την μου, από συνάδελφό μου. Στην Ελλάδα μιλάμε πάρα πολύ για τις ψευδείς ειδήσει και για την, τον ηγετικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Πέρα από την ε, στρατηγική επικοινωνίας, όπου λέτε για το τι κάνει η Ευρώπη για αμάς, για όλους τους πολίτες. Είναι αμυντικό όπλο αυτή η στρατηγική για τους ηλικιωμένους, για διάφορες κατηγορίες πολιτών. Δεν ξέρω αν είναι το όπλο, αλλά είναι ένα όπλο. Και θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά που έχουμε. Είναι ένα από τα στοιχεία που και μία, ένα από τα όπλα μας είναι να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει. Ε, έχουμε και μία task force που έχουμε δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο μιλητής. Έχουμε 14-15 ανθρώπους που ασχολούνται με τα fake news, ε, ανήκουν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και μέσα από διάφορες ανοιχτές πηγές εξετάζουν τι συμβαίνει πού. Ποιος επιτίθεται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέτεια. Και έχουν κάθε φορά αναπτύξει ένα αφήγημα που καταρρύπτει αυτές τις ψευδείς ειδήσει. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο ένα κώδικα διοντολογίας έχουμε ετοιμάσει που την έχουμε στο Facebook, στο Instagram, στο Google, στο Twitter, στις μεγαλύτερες πλατφόρμες δηλαδή. Και σε αυτόν τον κώδικα διοντολογίας, σε εθελοντική βάση, οι πλατφόρμες αυτές, όταν κάποιος τους λέει ότι κάποια πληροφορία είναι ψεύτικη ας πούμε, το τσεκάρουν και δέχονται να κατεβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη ψεύτικη είδηση από την πλατφόρμα. Είδαμε μια πρώτη έκθεση για το πώς λειτουργεί αυτός ο κώδικας διοντολογίας, πώς τα πάει στο facebook ας πούμε. 89% των αιτήσεων για να αφαιρεθεί μία ψευδής είδηση υλοποιήθηκε. Δηλαδή δόθηκε συνέχεια και κατέβηκε η είδηση. Επομένω είναι θετικό αυτό για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμόνο που ήρθε εδώ. Θα πρέπει να διάσουμε την αίθουσα, να καθαριστεί, γιατί στι 5 η ώρα ξεκινάει μία νέα συνεδρίαση. Σα παρακαλώ, ετοιμαστείτε για να βγείτε από την αίθουσα. Ευχαριστεί η Πρόεδρος και του Διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε και εμεί. Θα σα ξαναδούμε αύριο. Γεια σα. Γεια σας. Όσοι θέλετε να πάτε στο γραφείο τύπου και να δουλέψετε τρία τέταρτα πριν από το κοκτέιλ, ακολουθήστε τον Αντώνιο, που σας κάνει νόημα. Και όσοι θέλουν να πάνε κατευθείαν για το κοκτέιλ, ε, να πάνε μαζί με τη Σεσίλια. Θα σας τα ξαναδούμε αύριο. Γεια σας.